στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι θα σας διαβιβαστούν όλα αυτά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο ίδιος κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και επίσης πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης ε, ε τυχών τροπολογιών ολοκληρώνεται απόψε στις 7. Η δε ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 9 το πρωί, στην αρχή της συνεδρίασης. Σας εύχομαι Καλό σας βράδυ και ε, τη διακοπή της συνεδρίας.